τότε ως προς την άσκηση του λειτουργήματος αυτού. Σας καλωσορίσω λοιπόν. Ο κύριος Σεριμπή επίσης μου ανακοίνωσε ότι έχει προσχωρήσει στην ομάδα των Πρασίνων. Οι αρμόδιες αρχές της Ουγγαρίας μου ανακοίνωσαν την εκλογή του κυρίου Ερικ